Good morning everybody. Καλημέρα σας. Αρχίζει η, μερίσια ε, η Ολομέλεια, η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση της κυρίας Νικόλ Κιλ για τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή. Έχετε τέσσερα λεπτά κυρία Συγήτρια. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους